task force από εδώ από τις Βρυξέλλες στις διαδικασίες αυτές τις εκλογικές. Στηρίξαμε επίσης και διάφορα κοινοβούλια ανά τον κόσμο, όχι μόνο δηλαδή τις κυβερνήσεις αλλά και τα κοινοβουλευτικά σώματα. Κάτι το οποίο βέβαια εσείς το καταλαβαίνετε από πρώτο χέρι εννοείται. Δώσαμε επίσης στήριξη σε ένα στα τρία κοινοβούλια ανά τον κόσμο. Ένα στα τρία κοινοβούλια ανά τον κόσμο δηλαδή πήρε βοήθεια από εμά. Μέσω τη συνεργασία αυτή επίση δώσαμε αρρωγή στην Αφρική, Αραβικέ χώρε, Ασία και σε θεσμικό επίπεδο για μεταρρυθμίσει στο θεσμικό τομέα, στη διοίκηση και επίση καταλήξαμε να βοηθήσουμε και στην ε, σύνταξη προγραμμάτων που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων κλιματικές αλλαγές και προστασία του περιβάλλοντος. Επίσης βοηθήσαμε χώρες που κινδυνεύουν από κρίσεις. Πολύ βασικός τομέας αυτός για μας. Άρα θέλουμε τη μείωση του κινδύνου για καταστροφές και βέβαια ανάκαμψη και ανακούφιση εφόσον υπάρχει μια τέτοια κρίση. Βοηθήσαμε 70 χώρες τα τελευταία αυτά χρόνια, από τις οποίες 30 είναι ευάλωτες χώρες. Στον τομέα λοιπόν της μείωσης των επιπτώσεων από φυσικές καταστροφές βοηθήσαμε Καζακστάν, Νεπάλ και άλλες χώρες να υιοθετήσουν μέτρα ώστε να είναι καλύτερα προετοιμασμένες σε περίπτωση που υπάρξει νέα φυσική καταστροφή, να μπορέσουν να αντέξουν περισσότερο εφόσον υπάρξει στο μέλλον μία κάποια καταστροφή και να προκληθούν λιγότερες υλικέ ζημιές. Ας πάρουμε σαν παράδειγμα το Πακιστάν, για να είμαστε πιο συγκεκριμένοι. Μετά τις πλημμύρες το 2010 στο Πακιστάν, βοηθήσαμε 5,5 εκατομμύρια ε, άτομα για να έχουν νέα κτίρια με μεγαλύτερη αντοχή, να ανακτήσουν τα περιουσιακά τους στοιχεία. 40% των ανθρώπων που βοηθήσαμε ήταν γυναίκες. Και αυτός είναι ο κανόνας στα προγράμματά μας για την απασχόληση μετά από τέτοιου είδου καταστροφές. Στις προσπάθειες ανάκαμψης δηλαδή 40% στόχος μας είναι οι γυναίκες. Η εταιρική αυτή σχέση μεταξύ μας επίσης βοήθησε να καλύψουμε διάφορα κενά ανάμεσα στην ανακούφιση και την ανάπτυξη. Θέτουμε δηλαδή τα θεμέλια για η φόρα ανάπτυξη. Όσο γίνεται πιο γρήγορα δηλαδή ξεκινάει το ανθρωπιστικό έργο. Δυστυχώ, ξέρετε, πριν υπήρχε αυτή η διχοτομία. Είχαμε την ανθρωπιστική βοήθεια από τη μια και την γρήγορη ανάκαμψη. Τώρα αυτό το χάσμα καλύπτεται και είμαστε πολύ πιο αποτελεσματικοί επιτόπου. Ξέρουμε δηλαδή ότι οι ανθρωπιστικές βοήθειες και η προσπάθεια που γίνεται για γρήγορη ανάκαμψη είναι πράγματα που πάνε χέρι-χέρι, πρέπει να γίνονται εκ παραλίλου. Αλλιώς δεν είμαστε αποτελεσματικοί και δεν καταφέρουμε να προσφέρουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε με την ανθρωπιστική βοήθεια. Γι' αυτό θέλουμε πιο γρήγορα να περνάμε και στο στάδιο αυτό της ανάκαμψης. Να αναφέρω επίσης και τη σημασία ε, που είχε η βοήθεια των, τον ε, αναπτυξιακού προγράμματος στο ΟΗΕ. Γιατί, κοιτάξτε, δεν είναι ότι εμείς πάμε και φεύγουμε. Όχι. Είμαστε εκεί. Μονίμως μένουμε στις χώρες αυτές που έχουν πληγεί για να είμαστε ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στην ανθρωπιστική βοήθεια και την ανάκαμψη. Η εταιρική σχέση λοιπόν είναι κάτι πολύ σημαντικό και ήταν πάρα πολύ σημαντικό και όσον αφορά την απάλληψη της ένδυας. Συνεργαζόμαστε λοιπόν μαζί σε διάφορες χώρες και έχουμε βοηθήσει πάρα πολλές χώρες για την απάλληψη της φτώχειας, σε συνεργασία μαζί σας βέβαια, με ένα πρόγραμμα μεταξύ άλλων που έχει να κάνει με τις αλλαγές στο κλίμα. Εδώ ξέρετε δραστηριοποιούμεθα και στις ανατολικές ευρωπαϊκές χώρες για την ε, μείωση του διοξιδίου του άνθρακα με μείωση 170.000 το χρόνο. Στην έκθεσή μας δείχνουμε ότι η συνεργασία μεταξύ μας ήταν πολύ σημαντική και οδήγησε σε πρόοδο ανά τον κόσμο. Τώρα βέβαια τι μένει να κάνουμε τι πρέπει να κάνουμε για να πάνε καλύτερα τα πράγματα στο μέλλον ακόμα. Και αυτό είναι επίσης ένα τμήμα της έκθεσης και πολύ γρήγορα θα αναφερθώ σε τέσσερις τομείς στους οποίους πιστεύω ότι μπορούμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα με την εταιρική σχέση μεταξύ μας. Ο πρώτος τομέας είναι η αναπτυξιακή ατζέντα μετά το 2015 και πώς θα συνεργαστούμε και θα προβληματιστούμε για το μέλλον και για τις εξελίξεις σε ένα κόσμο που σίγουρα θα συνεχίσει να αλλάζει και θα αλλάξει άρα και η μελλοντική μας συνεργασία. Δεύτερον, μείωση της ένδυας και στόχοι της χιλιετίας. Πώς θα συντεριαστούν καλύτερα με τις κλιματικές αλλαγές και την προστασία του περιβάλλοντος. Γιατί είναι αλήθεια ότι έχουμε από τη μια μεριά την ένδυα και από την άλλη μεριά την προστασία του περιβάλλοντος και τις κλιματικές αλλαγές. Μιλάμε για την εφόρο ανάπτυξη. Λοιπόν, όταν όσοι ασχολούνται με την ένδια ε, συζητούν, τι λένε, λένε ναι, πρέπει να στηρίξουμε και τους άλλους στόχου, αλλά προτεραιότητά μας είναι ένδια. Και όταν μιλάτε με τους άλλους που ασχολούνται με την περιβάλλον, λένε θέλουμε αηφόρα ανάπτυξη, ναι, αλλά η κύρια διάσταση πρέπει να είναι το περιβάλλον. Οπότε εμείς στον ΟΙΕ πιστεύουμε ότι αυτά τα δύο πρέπει να συνδυαστούν, να βρούμε τη χρυσή τομή μεταξύ τους και να λειτουργήσουμε αλλιώς το μέλλον. Ειλικρινά πιστεύω ότι πρέπει να σταματήσουμε να μιλάμε για τα trade-offs και πρέπει να μιλάμε για μια σχέση από που όλοι να βγαίνουν κερδισμένοι. Αλλιώς θα βρισκόμαστε σε αντιπαράθεση μεταξύ μας και δεν θα καταφέρουμε να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε επιτόπου, ώστε να έχουμε ανάπτυξη με συνοχή και που να καλύπτει όλους, προκειμένου και να παλύψουμε τη φτώχεια και να πετύχουμε την προστασία ε, του περιβάλλοντος, γιατί αυτό είναι η αηφόρος ανάπτυξη και τα δύο. Ξέρουμε πώς να μιλάμε για αυτά, αλλά δεν ξέρουμε πώς να τα συνδυάσουμε καλύτερα επιτόπου. Ξέρετε, κατά πάσα πιθανότητα, γιατί, γιατί και τα χρήματα είναι κάπως χωρισμένα. Σημασία δεν έχει το από πού θα έρθουν τα χρήματα και πού ακριβώς θα βρεθούν. Οι στόχοι πρέπει να επιτευχθούν. Το δεύτερο θέμα που θα μας απασχολήσει είναι η ενέργεια. Η πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα όσον αφορά την ενέργεια για όλους είναι κάτι που θα μας απασχολήσει στο μέλλον. Και το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΟΗΕ έχει τοποθετηθεί όσον αφορά τις λύσεις για την ενέργεια, τα ενεργειακά δίκτυα, πώς θα βοηθήσουν τους πιο φτωχούς. Ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί είναι η ισότητα μεταξύ των δύο φύλων. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να ενισχύσουμε τις γυναίκες και να κάνουμε περισσότερα μαζί σας, σε συνεργασία μαζί σας για να το πετύχουμε αυτό. Και τέλος, μείωση των, φυσικών, ε, των επιπτώσεων των φυσικών καταστροφών και ανάκαμψη μετά από τις κρίσεις. Εδώ σημασία έχει τοπική δίκηση. Δημοκρατική δίκηση φυσικά και διακυβέρνηση. Για να πετύχει αυτό πρέπει να ενισχύσουμε την τοπική διάσταση. Τέλος, θέλω να υπογραμμίσω ότι η έκθεση που σας παρουσιάζουμε σήμερα δείχνει πώς η εταιρική σχέση μεταξύ μας έχει προχωρήσει, έχει κάνει τον κόσμο καλύτερο, έχει κάνει τη διαφορά. Είναι μια ιστορία επιτυχίας, μια αισιόδοξη ιστορία όπως είπατε κι εσείς. Τώρα πρέπει να στραφούμε στο μέλλον, να συζητήσουμε πώς θα διασφαλίσουμε την εξέλιξη της εταιρικής αυτής σχέσης. Έτσι, ώστε να συνεχίσει να είναι αποτελεσματική και να επηρεάσει τους επόμενους στόχους μας για να παλευθεί η ένδια και να πετύχουν οι στόχοι της εφόρου ανάπτυξης. Τέλος, ευχαριστώ πολύ τον Αντώνιο Φιχιλάντε. Αντώνιο, πραγματικά έχει βοηθήσει πάρα πολύ να βοηθήσω όλη την ομάδα του αναπτυξιακού προγράμματος του ΟΙΕ, UNDP, και όλους όσοι συνεργάστηκαν από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να πετύχει η προσπάθεια αυτή. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you. very Ευχαριστώ πάρα πολύ Ρεβέκα. Από το 2004 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δώσει 2,4 ευρώ για τις ενέργειες της UNDP του αναπτυξιακού προγράμματος του ΟΗΕ με κύριους ε, αποδέκτες το Ιράκ και το Αφγανιστάν 400.000 ευρώ και παραπάνω για κάθε μία από αυτές τις χώρες και συνέχεια η Νιγηρία και το Μπαγκλαντές. Υπάρχει λοιπόν αυτή η εταιρική σχέση για την πρόληψη των κρίσεων και των συγκρούσεων. Κύριε τι Τιμάλο, θα ήθελα να ακούσω από τα δικά σας χείλη κατά πόσο θεωρείτε ότι η UNDP, το αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΟΗΕ, έχει ένα συγκριτικό πλεονέκτημα ή αν και άλλοι εταίροι μπορούν να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα. Κύριε Ντιμέλο, να σας ε, θέσω ακόμα ένα ερώτημα. Βλέπετε κάποια ανάγκη να τροποποιηθεί αυτή η εταιρική σχέση, να θεσπίσουμε νέες προτεραιότητες για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε καλύτερα στο θεματολόγιο ανάπτυξης μετά από το 2015. Η Ρεβέκα μας έθεσε και μία πρόκληση. Είπε ότι η UNDP μπορεί να αντιμετωπίσει τα θέματα της εξάλληψης της ε, ένδυας και της βιώσιμης ανάπτυξης μέσω του κλιματικού θεματολογίου για το οποίο υπήρξε μια υπόσχεση για ένα δισεκατομμύριο ευρώ, αλλά δεν βλέπω τα χρήματα αυτά να έχουν δοθεί. Πώς μπορούμε λοιπόν να υλοποιήσουμε τις ε, υποσχέσεις μας, να προστατεύσουμε τις πιο τροτές χώρες, τις πιο τροτές αναπτυσσόμενες χώρες από την κλιματική αλλαγή. Και η χώρα από την οποία προέρχομαι είναι μια χώρα η οποία βρίσκεται εν μέρη κάτω από το νερό και βυτίζεται όλο και περισσότερο. Πώς προστατεύει κανείς τις χώρες αυτές από τη σημαντική αυτή απειλή που προέρχεται από την κλιματική αλλαγή. Δεν βλέπω να υπάρχει χρηματοδότηση ιδιαίτερη σε αυτό το τομέα και για την ε, αντιμετώπιση της ένδυας. Γι' αυτό η δική μου επιτροπή τουλάχιστον θεωρεί ότι δεν έχει νόημα να πάρουμε χρήματα από την ε, αντιμετώπιση τωρινών αναγκών για να περάσουμε στην, ε, ε, στο μετριασμό των ε, επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Αλλά ήταν ενδιαφέροντα αυτά που είπε η Ρεμπέκα. Κύριος Δημιαλό. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε θα κάνω μερικές σύντομες παρατηρήσεις προσπαθώντας να αντιμετωπίσω το θέμα αυτό το οποίο θέσατε εσείς ο ίδιος. Ε, κυρία Γκρίστον, ε, κύριε Πρόεδρε, έντιμο μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θέλω καταρχήν να ευχαριστήσω το πρόγραμμα ανάπτυξη των ΗΠΑ για τις προσπάθειες που έχει ε, καταβάλει και τώρα ε, χαιρετίζουμε και γιορτάζουμε τα 10 χρόνια τη εταιρική μας σχέση. Η έκθεση που παρουσιάστηκε από τη Ρεμπέκα είναι μια ε, συνολική επισκόπηση τη κοινή μα εργασία ξεκίνησε με την υπογραφή το 2004 μιας συμφωνίας εταιρική σχέσης και στη συνέχεια μπορούμε να δούμε ότι ακολούθησε μια δεκαετία σημαντικών επιτεύξεων. Πρώτα απ' όλα να υπογραμμίσω τη σημασία του να λειτουργήσουμε από κοινού μέσα σε ένα πολιτικό διάλογο. Η εταιρική μας σχέση λειτουργεί θετικά γιατί έχουμε μία εμπροστόστροφη αντιμετώπιση και θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις μεροδικές προκλήσεις. Το UNDP, το πρόγραμμα ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, είναι ένας εταίρο με τον οποίο μπορούμε να συζητήσουμε όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ανάπτυξη. Μια τέτοια συνεργατική προσέγγιση βοηθάει την προσπάθειά μας για να θεσπίσουμε τους στόχους ανάπτυξης επέκεινα του 2015. Πιστεύουμε ότι η αντιμετώπιση της ε, ένδυας θα πρέπει να συμβαδίζει και με άλλες ενέργειες με τη δημιουργία ενός πλαισίου το οποίο θα είναι πρόσφορο σε μια γενική εταιρική σχέση που να συνενώνει διεθνείς οργανισμούς, κοινωνία των πολιτών και πολίτες από όλες τις χώρες της γης. Βλέπουμε λοιπόν τη δυνατότητα να υπάρξει η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της UNDP επί τη βάση αυτών των ε, προτάσεων και συστάσεων που θα ενθαρρύνουν τον πολιτικό διάλογο και την κοινή δράση. Κατά την άποψή μου, κύριε Πρόεδρε, για τα θέματα των πόρων που θα πρέπει να δοθούν, θα πρέπει να απαντηθεί αυτό το ερώτημα με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων. Δεν θεωρούμε ότι η παραδοσιακή κυβερνητική αρρωγή για την ανάπτυξη πρέπει να είναι η μόνη λύση. Θα πρέπει να αναζητήσουμε και άλλες πηγές από εγχώριους πόρους ενδεχομένως, αλλά και τις, ε, τα εμβάσματα από τους εργαζόμενους που έχουν μεταναστεύσει από αυτές τις χώρες και επίσης και τη βοήθεια χρηματοπιστωτικών φορέων. Όλοι αυτοί οι πόροι λοιπόν θα πρέπει να εξεταστούν και να τεθούν στην υπηρεσία της ε, ανάπτυξης. Αλλιώς δεν νομίζω ότι μπορούμε να επιτύχουμε σημαντικά αποτελέσματα. Και στη διαδικασία επέκεινα του 2015 πιστεύω ότι διάφοροι εταίροι από διάφορες πλευρές του κόσμου θα πρέπει να συνεργαστούν δεδομένου ότι έχουν καταλήξει σε αντίστοιχα συμπεράσματα. Πριν από δύο μήνες στο Μεξικό συζητήσαμε τα θέματα αυτά και είδαμε όπως αντανακλάται και στο έγγραφό μας να υπάρχει μια γενική σύγκληση απόψεων ότι είναι απαραίτητο να κινητοποιήσουμε ένα ευρύτερο φάσμα πόρων για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα θέματα της ε, παγκόσμιας ανάπτυξης. Το σχέδιο του UNDP για το διάστημα 2014-2015 θέλει να αντιμετωπίσει την ένδια με τον αντιμετωπίσιμο ολοκληρωμένο τρόπο τα θέματα ανάπτυξης. Οι κύριες εστιακές περιοχές για το έργο στο νέο αυτό σχέδιο είναι η βιωσιμότητα, η αηφορία δηλαδή, η συμπερίληψη και η ανάπτυξη. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν μπορούμε να επιτύχουμε μια μεγαλύτερη βελτίωση της κατάστασης. Εδώ μεταξύ η συνεργασία μας ήδη αποφέρει καρπούς. Ιδίως σε σχέση με τους τρεις πυλώνες που βασίζεται η αντιμετώπιση μας. Ευκυβερνησία, αντιμετώπιση των συγκρούσεων, ανοικοδόμηση μετά τις συγκρούσεις. Η UNDP παίζει ένα σημαντικό ρόλο σε πολυμερές επίπεδο. Η συνεργασία μας δίδει εκλογική υποστήριξη σε πάρα πολλές χώρες που αναφέραμε προηγουμένως, κυρίως στις αφρικανικές χώρες. Στη Ζιμπάμπουε έχουμε συνεργαστεί για τη διαδικασία εκπόνησης ενός νέου συντάγματος. Χάρη στην κοινή αυτή προσπάθεια μπορούν οι πολίτες της Ζιμπάμπουε να ψηφίσουν όσον ούπο για ένα νέο σύνταγμα. Η εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως της Κομισιόν και της UNDP, είναι ιδιαίτερα προχωρημένη χάρη στο νομικό πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί και τη δυνατότητα συνεργασίας. Εμείς νομίζουμε ότι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε από κοινού τα παγκόσμια αυτά προβλήματα με πολυμερή υποστήριξη. Οι κοινέ μα για την αντιμετώπιση των ε, συγκρούσεων και την επίλυση των προβλημάτων ε, στέφθησαν με επιτυχία. Ε, δείτε την ακτή του ελεφαντοστού. Συνεργαστήκαμε με τη UNDP ώστε να ενισχύσουμε τα θεσμικά όργανα μετά από τη βία που ακολούθησε τις εκλογές του 2011. Επιπλέον στην Αγκόλα, στο Λίβανο, η δική μα συνεργασία στήριξε διάφορα πολυάριθμα προγράμματα και μπόρεσε να να βοηθήσει ώστε να αρθεί, ε, να, να αποναρκοθετηθούν τα, οι διάφορες περιοχές. Γι' αυτό τώρα μπορεί ο κόσμος να έχει πρόσβαση στα σχολεία αλλά και στα νοσοκομεία, αλλά και να ξεκινήσει ανοικοδόμηση. μπορούμε να κάνουμε διαφορά στον απλό κόσμο. Ε, πρόκειται για μια ισχυρή δύναμη για υπέρ της ειρήνης και της ανάπτυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στον κόσμο. Είμαστε βέβαιοι πως οι προσπάθειές μας θα ωφεληθούν περισσότερο από τον ε, ε, ενεργό και δραστήριο διάλογο. διακυβέρνηση, πρόληψη των κρίσεων και ανάκτηση μετά από την κρίση. Αυτό είναι μια καλή αναφορά γιατί προσπαθούμε να επιτύχουμε ταυτόχρονα και τους στόχους της χιλιετίας αλλά και να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε τη φτώχεια και να φτάσουμε περισσότερο, πιο εύκολα και πιο αποτελεσματικά στον κόσμο που το χρειάζεται. Ε, χρειάζεται να συνεχιστεί ο διάλογος για τα θέματα της βιώσιμης ανάπτυξης μέχρι το διεθνής διασκέψη του 2015. Σε διεθνές επίπεδο η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει μέσα στο πλαίσιο του 2015 και να, με οικοδομητική συνεργασία με την UNDP. Ε, χρειαζόμαστε ε, ε, να αντιμετωπίσουμε τις παγκόσμιες προκλήσεις με καθολική δράση. Μπορούμε να συνεργαστούμε για να δημιουργήσουμε συνέργειες και να έχουμε απτά αποτελέσματα και ουσιαστικά αποτελέσματα. Είναι και η ώρα να δούμε πώς από κοινού μετά από το 2015 θα μπορέσουμε να μετατρέψουμε την προσήλωσή μας σε στοχευμένη καλύτερα βοήθεια και να ε, ε, ε, κινηθούμε προς το όραμα μιας αξιοπρεπούς ζωής για όλους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ντιμέλο. Θέλω να προσκαλέσω τώρα τους συναδέλφους, αν θέλουν να λάβουν το λόγο. Σας παρακαλώ να περιοριστείτε σε δύο λεπτά. Γιατί είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θέλουν το, το λόγο. Ο Ρικάρδο πρώτος. Ο Ρικάρδο Κόρτες ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ τη Ρεμπέκα για την έλευση της στο Κοινοβούλιο και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να ξαναβρεθούμε σε σύντομο χρονικό διάστημα και θα διατηρηθεί αυτή η συνεργασία που έχουμε και θα ενισχυθεί περαιτέρω. Όλα φαίνεται να δείχνουν ότι οι νέες ευθύνες σου για την Λατινική Αμερική θα μας φέρουν πιο κοντά. Και θα ήθελα εδώ να αναφερθώ στο έργο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα θέματα τη Λατινική Αμερική. Ξέρετε ότι εμεί έχουμε εργαστεί ιδιαίτερα σε σχέση με την έκθεση που αφορά τι νέε μορφέ συνεργασία μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Λατινική Αμερική, μεταξύ των οποίων και το εργαλείο αυτό τη ανάπτυξη και συνεργασία με τον σοσιαλιστή εξεβονίμων μου ω εισηγητή. Ξέρετε λοιπόν ότι αυτό ενδιαφέρει ιδιαίτερα την Επιτροπή ανάπτυξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και το Συμβούλιο έχει μόλις αποφασίσει να δώσει μια συνέχεια στο αίτημα της ομάδας μου να αναβαθμιστούν οι σχέσεις μας με την Κούβα. Θέλουμε λοιπόν να έχουμε αυτήν <clears throat> την ε, νέα αντιμετώπιση των ε, χωρών της Λατινικής Αμερικής που εστιάζει και στις φτωχές χώρες αλλά και στις χώρες μέσου εισοδήματος. Εκεί βρίσκονται τα 70% των φτωχών στον κόσμο. Έχουμε επίσης εξασφαλίσει να υπάρχει ένας κανονισμός για τη συνεργασία που έχει σαν στόχο την εξάλληψη της ε, ένδυας αλλά και της ανισότητας με συνεργασία με ΜΚΟ επιτόπου στη Λατινική Αμερική. Ξέρετε λοιπόν, θα πρέπει να ξέρετε ότι είμαστε σύμμαχοί σας γιατί αυτή η περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μονάχα για την μεγάλη δημογραφική και οικονομική ανάπτυξή της, όχι για την διεθνή της θέση που την έχει κάνει ένα σημαντικό εταίρο και σύμμαχο σε παγκόσμιο επίπεδο, για τον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής ή τον έλεγχο των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θέλει να συνεχίσει να αγωνίζεται στον αγώνα κατά της ε, ε ανισότητος υπέρ της ε, κοινωνικής δικαιοσύνης και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπως είναι στην Κολομβία για την εδραίωση ειρενευτικών διαδικασιών. Ένα απλό ερώτημα μονάχα θέλω να θέσω. Ποιο πώς βλέπετε αυτόν το ρόλο της Λατινικής Αμερικής για, την καλύτερη, τον καλύτερο προσδιορισμό των στόχων της ανάπτυξης μετά από το 2015 και ποιες είναι οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Λατινική Αμερική και ποιος θα πρέπει να είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής και είναι η ευκαιρία η παρουσία του κ. Φρουτουόζου για να μας απαντήσει και αυτός εάν θέλει. Χωρίς μικρόφωνο ο πρόεδρος, ο κύριος Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ. Και εγώ θέλω να καλωσορίσω τη Ρεμπέκα Κρίνσπαν, γιατί είναι, και θα τη συγχαρώ φυσικά για τα εξαιρετικά αποτελέσματα που έχει επιτύχει ε, από τη στιγμή που ανέλαβε τα ηνία αυτού του προγράμματος ανάπτυξης. Νομίζω ότι η συνεργασία αυτή ε, με την Κομισιόν και τον κύριο ως Δεμέλο, θα μπορούσε, κάνοντας ένα λογοπαίγνιο στο όνομά του, να πω ότι ήταν ιδιαίτερα καρποφόρα. Η ανάπτυξη στόχων πέρα από το 2015, ε, μετά από το 2002 που τέθηκε σε εφαρμογή αυτό το πρόγραμμα, έχουμε μειώσει κατά 5 εκατομμύρια τον αριθμό των πτωχών, έχει μειωθεί κατά 30% η παιδική και τα 25% τα κρούσματα ελαιονοσίας. Τώρα όμως πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους στόχους πέραν του 2015 και φυσικά έχουν αλλάξει τα πράγματα διότι ο παγκόσμιος πληθυσμός έχει αυξηθεί κατά ένα δισεκατομμύριο και παραπάνω. Έχουμε νέους παίκτες στο παγκόσμιο χώρο και όπως είπε και η κυρία Γκρίνσπαν είναι απαραίτητο να συνδέσουμε τους στόχους μείωσης της ένδυας με τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτή λοιπόν η αλλαγή αντιμετώπιση που παρουσιάζεται στον ΟΗΕ παρουσιάστηκε μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πολλά κρατημέλη που θέλουν να δώσουν μεγαλύτερη έμφαση στα θέματα αυτά. Εγώ θα ήθελα να ξέρω σε ποιο βαθμό μετά από τη συνάντηση του Ρίο, όπου θεσπίστηκαν τα στοιχεία της βιώσιμης ανάπτυξης, πόσο μπορούν, σε ποιο βαθμό μπορούν να τροποποιηθούν αυτοί οι στόχοι και δύο ερωτήματα. Πρώτο, σε ποιο βαθμό οι υποβόσκουσες συγκρούσεις είναι το κυριότερο πρόβλημα για να μπορέσουν να επιτευχθούν οι στόχοι του, της χιλιατίας και σε δεύτερο βαθμό πόσο μπορεί να συμπεριληφθεί και το θέμα της εργασίας, γιατί ο Παγκόσμιος Οργανισμός Εργασίας ουσιαστικά είναι στο περιθώριο των στόχων της χιλιετίας, αλλά το γεγονός ότι υπάρχουν προβλήματα με την άτυπη εργασία, με τις συμπίε των μισθών και όλα αυτά. Όλα αυτά είναι θέματα τα οποία έχουν επίπτωση στα ζητήματα αυτά. Και ως πρόεδρος της Επιτροπής ε, Ευρωλάτ, τη αντιπροσωπεία τη Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ευρωλάτ, έχουμε υποστηρίξει ιδιαίτερα τι προσπάθειε του κυρίου Μπέρμαν και του κυρίου Κορτέ Λάστρα, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι η Λατινική Αμερική θα μπορέσει να συμμετάσχει περισσότερο στην επιτεύξη των στόχων αυτών τη ανάπτυξη και η ελπίδα μα είναι ότι η Κομισιόν θα μπορέσει και αυτή να κάνει τι απαραίτητε προσπάθειε και να μα βοηθήσει ώστε να συνεχίσουμε να βοηθούμε τι χώρε τη Λατινική Αμερική με την χρηματοδότηση αυτή. Ευχαριστώ. Ε, Ευχαριστώ πολύ και τον κύριο Κορτές και τον κύριο Σαλαφράγκα για τα όσα είπατε. Κοιτάξτε, σήμερα το απόγευμα προβληματιζόμαστε για τα αποτελέσματα του προγράμματός μας και για το μέλλον του. Ο κόσμος δεν θα καταφέρει να αντιμετωπίσει τα προβλήματα της κλιματικής αλλαγής ή της αηφόρου ανάπτυξης αποκλείοντας τις χώρες αυτές μέσου εισοδήματος. Οι στόχοι μας όσον αφορά τις κλιματικές αλλαγές και την αηφόρο ανάπτυξη θα επιτευχθούν μόνο μαζί με αυτές τις χώρες και όχι χωρίς αυτές. Συνεπώς, το θέμα είναι πώς θα συμμετάσχουν στην προσπάθεια αυτή και θα διδούν σε μια συνολική, συλλογική προσπάθεια και όχι σαν μια προσπάθεια τοπική. Το θέμα της χρηματοδότησης για την ανάπτυξη είναι κάτι που πάει πολύ πιο πέρα από το θέμα της αρρωγής. Δεν είναι το μόνο μέσο εξάλλου για την διεθνή συνεργασία για την ανάπτυξη. Χρειάζεται λοιπόν μεγαλύτερη συμμετοχή σε αυτό που ονομάζουμε συνεργασία νότου-νότου στον τομέα της έρευνας, της γνώσης, της εμπειρίας. Αλλά υπάρχει και ένα δεύτερο στοιχείο. Και αυτό είναι ότι δεν θα υπάρχει εφόρος ανάπτυξη αν αποκλείσουμε τον ιδιωτικό τομέα από τις προσπάθειές μας. Οι χώρες αυτές λοιπόν μέσου εισοδήματος είναι αυτές που πρέπει να συμμετάσχουν με τον ιδιωτικό τομέα, με τις κυβερνητικές οργανώσεις, προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα των κλιματικών αλλαγών και της αηφόρου ανάπτυξης. Δεν είναι θέμα αρρωγής. Μιλάμε για χρηματοδότηση για την ανάπτυξη που σημαίνει επίτευξη των στόχων μας που είναι η αηφόρος ανάπτυξη και η αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών με τις χώρες αυτές. Γιατί αλλιώς ξεκινάμε με αποτυχία βεβαιωμένη. Οι χώρες αυτές είναι μέρος της λύσης και όχι του προβλήματος. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ξέρουμε για να προσαρμόσουμε ανάλογα τους στόχους μας. Βλέπετε, από τη δεξινόμηση της Παγκόσμιας Τράπεζας υπάρχουν οι φτωχές χώρες, οι μεσαίες και εκείνες υψηλών εισοδημάτων. Και τι μένει τελικά. Όλες οι χώρες έχουν ε, ανέβει. Και γι' αυτό και οι χώρες που είχαν πολύ χαμηλό εισόδημα τώρα έχουν ε, περάσει περισσότερες τουλάχιστον στην πιο πάνω κατηγορία, μέσων εισοδημάτων. Τα τελευταία 15 χρόνια έχει γίνει αυτή η αλλαγή, 20. Οπότε πρέπει να αναρωτηθούμε, οπότε τελικά τι νόημα έχουν αυτές οι κατηγορίες, εφόσον οι χώρες αυτές μέσους δεν τι είναι. Είναι από το πράσινο ακροτήρι μέχρι την Αργεντινή. Κατά κάποιο τρόπο δηλαδή, και αυτό ρώτησε και ο Γνάθιο Σαλαφράγκα, πρέπει να μιλήσουμε για το βαθμό στον οποίο είναι τρωτή μια χώρα. Υπάρχουν χώρες που βρίσκονται συνεχώς σε κρίση, σε συγκρούσεις ανά τον κόσμο. Και έρχομαι στο τελευταίο. Δεν μπορώ να τα απαντήσω όλα βέβαια, αλλά θέλω να κάνω την εξής παρατήρηση. Δεν θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την ένδια αν δεν έχουμε αν δεν αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο κάνουμε τα πράγματα στο μέλλον. Πρέπει να αλλάξουμε. Ένα στοιχείο θα σας δώσω και θα τελειώσω με αυτό. Ο κόσμος που ζει από τα οικοσυστήματα είναι 2 εκατομμύρια στον κόσμο που ζουν δύο δις άνθρωποι. Άρα πρέπει να προσαρμόσουμε την πολιτική μας, να στηρίξουμε τα οικοσυστήματα, αυτά που είναι πιο τροτά, πιο ευάλωτα, για να μπορέσουμε να στηρίξουμε αυτά τα δύο δισεκατομμύρια ανθρώπους. Πώς θα απασχοληθούν οι άνθρωποι αυτοί, δεν θα υπάρχουν αρκετές θέσεις απασχόλησης για να απασχοληθούν αυτοί. Και εκεί είναι που συνδυάζονται η φτώχεια με το περιβάλλον. Αν δεν το κάνουμε αυτό, οι προσπάθειές μας θα αποτύχουν. Κοιτάξτε, ο χρόνος ε, τρέχει και ήθελα απλά να πω ε, ότι πρόσφατα ε, ακούσαμε ότι το Δελχή είναι η πιο μολυσμένη πόλη του κόσμου και πρόκειται για μια χώρα με μέσο εισόδημα, ενώ το Μπαγκλαντές που είναι πιο φτωχή χώρα, είναι πιο βιώσιμη όσον αφορά τις, τις κλιματικές αλλαγές. Ενώ μια μέσο εισοδήματος χώρα δεν μπορεί να τα καταφέρει. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Λοιπόν, και τώρα ο Τζο Λάινεν έχει ζητήσει το λόγο και ο Μιγγέλ Μαρτίνες. Κοιτάξτε, εγώ δεν θέλω να κάνω παρουσίαση, αλλά να εισήγηση, αλλά να θέσω μια ερώτηση. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε. Είχα τη χαρά να σας συναντήσω και ήρθαμε μια προσωπία και στη Νέα Υόρκη. Ε, το πρόβλημα της εποχής μας τα επόμενα 20, 30 έως και 50 χρόνια είναι το να τραβήξουμε το κοινό κοντά μας. Ωραία, ε, ένα περισσότερο με το ίντερνετ και την αραβική άνοιξη κτλ. Πρέπει να έχουμε τη στήριξη του κοινού και να το παρασύρουμε. Αυτό ισχύει για τις κλιματικές αλλαγές, για τους στόχους της ανάπτυξης και για όλα με όσα ασχολούμαστε εμείς οι πολιτικοί. Στη χώρα μου, το Ηνωμένο Βασίλειο, υπάρχει μια αυξανόμενη ε, ε, κίνηση από τις φρικτές ε, εθνικές ε, εφημερίδες ε, τις χρησιμοποιούν μόνο για να φτιάχνουν αναχώματα για τις πλημμύρες ε, πια. εσύ τι μπορείς να κάνεις Ρεβέκα για να πουλήσεις αυτές τις ιδέες σου στον κόσμο. Εμείς εδώ τις συμμεριζόμαστε όχι μόνο στη δική μου χώρα αλλά γενικά σε όλους. Να προσπαθήσουμε δηλαδή να γνωστοποιήσουμε τα τι κάνουμε, να φτάσουμε στον κόσμο. Δεν ε, αρκεί πια το να περνά από κυβερνήσει κοινοβούλια κτλ. Εσεί, τι θα κάνετε γι' αυτό λοιπόν. Ευχαριστώ. Τώρα για ποια χώρα μιλά εσύ. Δεν μιλάς για την Μεγάλη Βρετανία. Ε, ο Τζορ Λάινεν. Καλώ όρισε, Ρεβέκα. Είναι εντυπωσιακό να βλέπουμε τα θέματα συνεργασίας μας σε πόσο μεγάλο φάσμα καλύπτουν εσύ είπες ότι το θέμα του κλίματος είναι σχετικά νέο, ωστόσο καλύπτει ένα μεγάλο τμήμα της εισήγησή σου ε, και συμφωνούμε πως θα αποκτήσει ακόμα μεγαλύτερη σημασία στο μέλλον, βιώσιμη ανάπτυξη στους τρεις πυλώνες της και μιλάμε συχνά για την τεχνολο... μεταφορά τεχνολογίας από εμά προς εκείνους ε, και εν μέρη αυτό είναι μάλλον απαραίτητο, αλλά υπάρχουν ε, τεχνολογίες που χρειάζεται να τις γνωρίσουν αυτοί οι λαοί, αυτά τα δύο δις που ζουν από τα περιβάλλον, να μπορέσουν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, ώστε να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τους πόρους που βρίσκουν και να ε, υπάρξει προστεθέμενη αξία για την οικονομία, αλλά και βέβαια και για τη βελτίωση της κοινωνικής τους κατάστασης. Εγώ θα ήθελα να δω λοιπόν πώς στη συνεργασία μας μπορούμε να εστιάσουμε στις τοπικές ε, δυνατότητες ώστε να βελτιωθούν τα πράγματα. Ευχαριστώ πολύ για αυτή την ε, συμβολή. Μαρτίνες, Μαρτίν. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θέλω να καλωσορίσω και την Ρεβέκα, αλλά και τους άλλους συναδέλφους που είναι εδώ. Κάθε φορά που μιλάμε με την Ρεβέκα, διαπιστώνουμε ότι η Ρεβέκα είναι πραγματικά μεγάλη πηγή έμπνευση. Και βέβαια είναι πολύ καλό πέρα από, τα... από την ίδια την προσωπικότητα της Ρεβέκας. Επιπλέον υπάρχει και το γεγονό της προέλευσής της, από πού έρχεται, πώς έχει ξεκινήσει στην πολιτική, στη χώρα της κλπ. κλπ. Πραγματικά νιώθουμε περήφανοι γι' αυτό. Φυσικά, όπως και οι συνάδελφοι που μίλησαν πριν από μένα, και εγώ χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να συνεχίσει να συνεργάζεται, όπως το έκανε μέχρι τώρα, στη σχέση αυτή και θέλουμε και εμείς να ενισχύσουμε το έργο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και γενικά η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσει να συνεργάζεται με τον ΟΗΕ. Και είναι καλό αυτό που ακούσαμε να λες, ότι είναι αποφασιστική σημασία η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ωραία. Σήμερα έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα να γιορτάσουμε. Θα συναντηθούμε με μη κυβερνητικέ οργανώσεις μετά από εδώ, που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα και θα συζητήσουμε μαζί τους το προεκλογικό πρόγραμμα εν ώψη των ευρωεκλογών. Και εφόσον υπάρχουν τέτοια αντίγραφα θα τους τα δώσω. Αν μπορούμε να έχουμε 10-20 τέτοια αντίτυπα να τους τα μοιράσουμε μετά. Τώρα, είμαι αντιπρόεδρος στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και είμαι υπεύθυνος για την πολυγλωσία. Μιλάμε όλες μας τις γλώσσες εδώ 24 ώρες το 24ωρο. Έτσι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να μας ακούνε στην γλώσσα τους. 80% των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση μιλάνε μόνο τη γλώσσα τους. Και μπορούν να μας ακούνε. Ό,τι τώρα συζητάμε εδώ πέρα, ο καθένας τα λέει στη γλώσσα του, ε, οι πολίτες μπορούν να το ακούσουν στη δικιά τους γλώσσα όλα αυτά. Και έτσι να νιώσουν ότι είναι δικό τους το θέμα που συζητάμε. Τι με απασχολεί εμένα τώρα με αυτό το έγγραφο. Το έγγραφο αυτό, αν υπάρχει σε μία μόνο γλώσσα, τότε 65% των ε, πολιτών μας δεν ενημερώνονται για το τι περιλαμβάνει, τι λέει. Και εμένα αυτό πραγματικά με νοιάζει. Θα ήθελα να κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε το έγγραφο αυτό να υπάρχει και στις υπόλοιπες γλώσσες, τέλος πάντων όσο γίνεται περισσότερες, ώστε να μπορούν να ενημερωθούν καλύτερα οι πολίτες. Γιατί κάποιοι ενδιαφέρονται. Και εξάλλου πρέπει να είναι κάτι γνωστό στους πολίτες, γιατί δεν είναι πολυτέλεια. Ό,τι περιλαμβάνει εδώ αυτό το έντυπο έχει πληρωθεί με τα χρήματα που βγαίνουν από την τσέπη των πολιτών. Νιούτον, αν οι Βρετανοί τα ξέραν αυτά, κανένας δεν θα πρότεινε να μην δαπανάμε σε αυτά. Και ένα τελευταίο. Κοιτάξτε, Το 70% των όσων βρισκόμαστε εδώ συμμετέχει στην ομάδα μας. Γιατί? Γιατί από την ταυτότητά του είναι η ομάδα εκείνη η οποία είναι πιο διεθνής και ενδιαφέρεται για τη συνεργασία στην ανάπτυξη. Γιατί είναι η ίδια φύση μας που μας οδηγεί σε αυτό. Και δεν το λέω σαν ε, μια ταμπέλα που μου βάζω, αλλά αντίθετα το λέω σαν δέσμευση που αναλαμβάνω να συνεχιστεί η συνεργασία αυτή μαζί σας. Να συνεχίσουμε λοιπόν στην πορεία αυτή εμβαθύνοντας, διευρύνοντας το πεδίο μας και έχοντας και νέες επιτυχίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Μιγγέλ. Έχουμε πίεση χρόνου όμω και επειδή πρέπει να απαντήσουν οι συνάδελφοι θα πρέπει να πιο σύντομοι αλλά έρχονται οι εκλογές βέβαια. Το βλέπω αυτό ο Νόρβετ. Ευχαριστώ πολύ. Προτιμώ να μιλήσω στα γερμανικά. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την ε, τόσο πλήρη και θετική έκθεση που μας έχετε παρουσιάσει σήμερα. Θα ήθελα από τη δική μου εμπειρία να παρατηρήσω ότι η συνεργασία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το πρόγραμμα ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, UNDP, λειτουργεί σωστά. Η συνεργασία λοιπόν της UNDP με την Ευρωπαϊκή Ένωση λειτουργεί θετικά. Είναι πάρα πολλά αναπτυσσόμενα κράτη τα οποία έχουν διαπιστώσει αυτή την πραγματικότητα. Αναφέρθηκε και Ζιμπάμπουε και εκεί είδα ποια είναι τα θετικά αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας. Αλλά δεν είναι τίποτα τόσο καλό ώστε να μην μπορεί να βελτιωθεί περαιτέρω. Και εγώ θέλω να θέσω ένα πιο αρνητικό παράδειγμα. Ρωτάμε για το μέλλον πώς μπορούμε να οργανώσουμε καλύτερα τη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Γιατί σε ορισμένες αναπτυσσόμενες χώρες υπάρχει η ανάγκη να ενισχύσουμε τις ε, ανανεώσιμες ενέργειες και την παραγωγή από εκεί. Και οι υπουργοί οικονομικών ή ενέργεια των χωρών αυτών μα, λένε πολλέ φορέ, με ποιον να διαπραγματευτούμε, με τα Ηνωμένα Έθνη, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχουμε κράτη τα οποία εργάζονται προς την κατεύθυνση αυτή, ΜΚΟ, οι Κινέζοι και αυτοί θέλουν ένα πόδι στην πόρτα. Το ερώτημα λοιπόν είναι πώς θέλουμε στο μέλλον να βελτιώσουμε αυτή τη συνεργασία και το συντονισμό ώστε να έχουμε τις απαραίτητε συνέργειες. Ένα δεύτερο σχόλιο έχει να κάνει με τους στόχους της χιλιετίας μετά από το 2015. Εδώ ένα σημαντικό στόχος είναι η βιώσιμη παραγωγή ενέργειας. Είναι από του μεγάλους στόχους του Ban Ki-moon. Πώς θεωρεί το UNDP μαζί με την Ευρωπαϊκή Ένωση να θεσπίσει αυτό το στόχο σαν ένα από τους κύριους στόχους της ε, χιλιετίας μετά από το 2015. Ευχαριστώ Νόρμπερτ. Η Άννα Γκάμις. Χαίρομαι πάρα πολύ Ρεβέκα όταν σε βλέπω κοντά μας. Ξέρεις ότι υποστηρίζω απόλυτα τον ρόλο των Ηνωμένων Εθνών. Πρέπει να πω όμως, απογοητεύομαι όλο και περισσότερο με πολλούς τρόπους με τους οποίους έχουμε από τη μια πλευρά μια εξαιρετική παρουσίαση στόχων, αλλά το αποτέλεσμα των συγκεκριμένων ενεργειών δεν βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο. Και αυτό αφορά και την UNDP και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι εδώ έχουμε ενώπιον μας ένα σημαντικό εγχείρημα. Ο Bill Newton Dunn μιλούσε για την πειθό που χρειάζεται έναντι της κοινή γνώμης, το να πείσουμε τους φορολογούμενους. Πιστεύω λοιπόν ότι πέραν της ε, πειθούς που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε προς την κοινή μας γνώμη και της αντιμετώπισης των αρνητικών αντιδραστικών κινήσεων που ανέφερε προηγουμένως, χρειαζόμαστε επιπλέον να πείσουμε την κοινή γνώμη στις χώρες όπου εργαζόμαστε και όχι μόνο τις δικές μας, εκεί που δαπανούμε τα χρήματα. Φοβάμαι λοιπόν, δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάνουμε πραγματικά όλα αυτά τα οποία μπορούν να περάσουν από το χέρι μας, αλλά δεν λαμβάνουμε υπόψη τα θέματα της ευκυβερνησίας, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες αυτές. Εγώ άνοιξα αυτό το βιβλίο και εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη περίπτωση που με ενδιαφέρει. Είδα να κάνετε θαύματα σε πολλές χώρες και φαίνεται αυτό και από τα, αυτά που περιγραφεί το έργο σας. Αλλά θέλω να αναφερθώ σε ένα συγκεκριμένο κράτος, την Αιθιοπία. Δεν οποιαδήποτε χώρα. Είναι η δεύτερη πιο πολυπληθής χώρα στην ε, Αφρική. Εκεί είναι η έδρα της Αφρικανικής ε, Ένωσης. Είναι ένας πραγματικός πελάτης βοήθειας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας από τους στόχους της δράσης της UNDP και αυτή η σελίδα που βλέπω εδώ πέρα είναι αποτροπιαστική γιατί δεν αναφέρει τίποτα για το ρόλο της κοινωνίας των πολιτών. Και φυσικά ε, υπάρχει νομοθεσία αυτή στην Αιθιοπία που ουσιαστικά απαγορεύει στην κοινωνία των πολιτών να αναπτύσσει την παραμικρή ενέργεια είτε είναι φιλανθρωπική είτε είναι υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Είναι πάρα πολλοί οι οποίοι είναι στη φυλακή, κυρίως δημοσιογράφοι. Δεν υπάρχει καμία αναφορά για το θέμα αυτό. Υπάρχει ένα πρόγραμμα αρπαγής γης στην Αιθιοπία που εμποδίζει τους ανθρώπους που ζουν ως γεωργοί στην Ήπεθρο να λειτουργήσουν και εδώ λέτε τι ωραία που είναι τα πράγματα στην Αιθιοπία. Αυτό με αποτροπιάζει, με ενοχλεί. Ο Τις Μπέρμαν. Ευχαριστώ πολύ. Ρεβέκα. Ζούμε στην καλύτερη δυνατή σφαίρα συνεργασίας μαζί σας. Ίσως θα μπορούσα να είμαι λιγάκι προκλητικός Θέλω να πάω σε μια συζήτηση τώρα σε λίγο για την ανάπτυξη και το μέλλον της ανάπτυξης από την ευρωπαϊκή πλευρά. Ίσως θα πρέπει να είμαστε όμως κάπως κριτικοί σε ορισμένα σημεία. Παρά το γεγονός ότι έχουμε τα εργαλεία για την αναπτυξική συνεργασία προσπαθούν να θεσπίσουν τις σωστές προτεραιότητες για την κλιματική αλλαγή, τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την περιεκτική ανάπτυξη, ίσως θα υπάρξουν κάποιες αλλαγές οι οποίες θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα ζητήματα αυτά. Και όλα αυτά περιστρέφονται γύρω στην δημοκρατική διαχείριση των σημαντικών προκλήσεων. Το πώς θα μπορέσουν να γίνουν καλύτερα, πώς να γίνει καλύτερα η κοινή χρήση των ε, φυσικών πόρων και θα έπρεπε να οργανώσουμε ίσως μια παγκόσμια ε, συνδιάσκεψη για το πώς μπορούμε να πετύχουμε κάθε χώρα να έχει το δίκαιο μεριδιό της. Πώς θα γίνει αυτό με έναν τρόπο που είναι δημοκρατικός. Νομίζετε ότι παίρνει αρκετέ πρωτοβουλίε η Ευρωπαϊκή Ένωση για τα θέματα αυτά. Εγώ νομίζω θα μπορούσαμε να κάνουμε και περισσότερα. Πρέπει οι φυσικοί πόροι να αντιμετωπίζονται με δημοκρατικό τρόπο. Υπέρ των πολιτών των χωρών αυτών. Και αυτά φυσικά περιλαμβάνουν και την ανακύκλωση, την ε, προστασία των ε, κύκλων παραγωγής από την αρχή ως το τέλος, νομίζω ότι έχετε τέτοια προβλήματα να αντιμετωπίσετε. Όσο πιο μεγάλη είναι η πυκνότητα του πληθυσμού, τόσο πιο προσεκτική πρέπει να είναι η ευκυβερνησία και η αντιμετώπιση όλων των εμπλεκομένων, ώστε ο καθένας να θεωρεί ότι σέβεται το σύστημα τα δικαιώματα και τις ανάγκες του. Οι ευμαρείς χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν κάποια καλή πείρα σε ό,τι αφορά αυτή τη λεγόμενη δημοκρατικού χαρακτήρα μηχανολογία σε ό,τι αφορά την επίτευξη της ευκυβερνησίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να βοηθήσει και τους άλλους. Πιστεύω ότι εδώ μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα στη δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και έχουμε από την άλλη πλευρά τα τροτά αυτά και εύθραυστα κράτη. Δεν νομίζω ότι κάνουμε αρκετά πράγματα για να έχουμε μια σωστή στρατηγική για τα εύθραυστα αυτά κράτη, όπως είχαμε ζητήσει το 2007-2008 και είναι φανερό ότι δεν υπήρξαν αρκετές προσπάθειες από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να έχετε μια πιο κριτική στάση για θέματα αυτά όπου μπορεί να έχετε μια πιο εχμηρή θέση. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και προβλέπαμε να το κάνουμε για μία ώρα το οποίο είναι βρωμοανεπαρκές. Συγγνώμη για για την ε,